γιατί αν δεν ενεργήσουμε τώρα θα σημειωθούν ακόμη σοβαρότερε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέλλον. Θα ήθελα να εμπλακεί λοιπόν πιο δραστηρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να παρακολουθήσει ε, την κατάσταση ω προ εκλογέ. Ευχαριστούμε. Ήσασταν τελευταία ομιλήτρια στα πλαίσια του, των παρεμβάσεων του άρθρου 150 και περνούμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση του κυρίου Φιλίδη. Ε, πρόκειται για την πολιτική προστασία των καταναλωτών. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε ε, το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών ότι θα παρουσιάσει την νέα πράξη για τα δικαιώματα των καταναλωτών τον Μάιο-Ιούνιο του 2012. Στη βάση αυτού, το Ευρωκοινοβούλιο ανάλαβε να συντάξει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για να βάλει το στίγμα του στη νέα πράξη. το σχέδιο έκθεσης αρχικά είχε αναλάβει εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας η εύα Βενσον, η οποία όμως αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει μετά την παραίτηση της για λόγους υγείας και μου ανατέθηκε να το ολοκληρώσω. εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην εύα Μπρίτ για την εργασία που πρόλαβε να κάνει σε αυτή την έκθεση και της εύχομαι να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούν τόσο η eva αρχικά αλλά και ο μιλών αργότερα θελήσαμε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και παραλήψεις του συστήματος και να περιλάβουμε πρόνοιες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών. βασική στόχη του σχεδίου έκθεσης όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρωταθέν προσχέδιο ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καταναλωτές η μείωση μέχρι και εξάλληψη των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των σχέσεων τους με τι εταιρείε, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών γενικά και με ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εναλλακτική επίλυση διαφορών η μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων και υψηλού επίπεδου προστασία των καταναλωτών η έμφαση στις ευπαθείς ομάδε του πληθυσμού με στόχο μια κοινωνικότερη ευρώπη καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας η οικολογία και η βιωσιμότητα η μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε επικίνδυνα χημικά όπως αντιβιωτικά στη βιομηχανία κρέατος τις παραβένες στα καλλιντικά μείωση των τεχνητών τρανσλιπαρών στα τρόφιμα η προστασία των παιδιών από τη διαφήμιση. όπως ήταν φυσικό κύριε πρόεδρε οι πιο πάνω στόχοι αντικρίστηκαν διαφορετικά από τις πολιτικές ομάδες που μέσα από 188 συνολικά τροπολογίες η κάθε μια πρότεινε τη δική της λύση στα διάφορα ζητήματα. σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν στην έκθεση όσες απόψεις ήταν δυνατό χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της έκθεσης διατυπώσαμε με τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών 16 συμβιβαστικές τροπολογίες και τελικά η έκθεση όπως διαμορφώθηκε τέθηκε σε ψηφοφορία στην επιτροπή εσωτερικής αγοράς στις 17 δεκάτου. υπερψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ 0 εναντίον και δέκα αποχές. ωστόσο το σχέδιο όπως ψηφίστηκε δεν άφηνε ικανοποιημένες ορισμένες πλευρές του κοινοβουλίου και αυτό γιατί ενώ επρόκειτο για μια έκθεση πάνω στη στρατηγική που αφορά τις πολιτικές για την προστασία του καταναλωτή αυτή ψηφίστηκε χωρίς την αναφορά στο στόχο για μια κοινωνικότερη ευρώπη ενώ διαγράφηκαν όλες σχεδόν οι αναφορές σε επικίνδυνα καρκινογόνα χημικά καθώς και η θέση για απαγόρευση της άμεσης τηλεοπτικής διαφήμισης που στοχεύει παιδιά κάτω των 12 ετών. Μετά από αυτή την εξέλιξη και ύστερα από συνεννόηση με όλες τις πολιτικές ομάδες, ανοίξαμε ένα νέο κύκλο συζητήσεων που οδήγησε τελικά στη δέσμευση όλων να στηριχθεί το προτινόμενο για ψήφιση αύριο συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές καθώς η οικονομική κρίση τους καθιστά πιο ευάλωτους, επιδιώκει μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων, τονίζει την ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ζητά υψηλό επίπεδο προστασία του καταναλωτή αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας εκφράζει ανησυχία για την εκτεταμένη διαφήμιση στην οποία εκτίθενται τα παιδιά και εισηγείται τρόπους καταπολέμησης της κατασπατάληση των τροφίμων θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν και τη σημαντικότατη προσφορά τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί συνένεση επί των βασικών πτυχών της έκθεσης και τη δέσμευσή τους για στήριξη της έκθεσης στην αυριανή ψηφοφορία. ευχαριστώ. Η δικασία catch the ε, ο κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή βάζει στο κέντρο της τους ε, καταναλωτές. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, αγαθών θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και όχι το αντίστροφο στην Ευρώπη υπάρχουν φοβερές διαιρέσεις και διχασμοί σε αυτό το λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλές προσπάθειες ούτω ώστε η πολιτική των καταναλωτών ε, από το 2002 να είναι υπέρ των καταναλωτών. Δημιούργησε δίκτυα καταναλωτών, ε, μίλησε ε, πολλές φορές για τη σημασία της πληροφόρησης, έκανε ενημερωτικές εκστρατείες για τους καταναλωτές, μελέτησε διάφορα προϊόντα. Ε, υπήρξαν διάφορες βέβαια παραβιάσεις, αλλά, αλλά έχουμε και τα εργαλεία πια για την προστασία όσων πέφτουν θύματα τέτοιων παραβιάσεων, προβλημάτων κτλ. Στη Σλοβακία ένα τμήμα δυστυχώς των παραγωγών δεν λαμβάνει υπόψη ε, τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών. Ελπίζω ότι οι κανόνες θα είναι πιο διαφανείς και καλύτερα εφαρμόσιμοι με βάση τη νέα πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών ε, είναι ατομικά δικαιώματα και γι' αυτό το λόγο πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, ε, πιο συγκεκριμένα τους καταναλωτές. Εξάλλου γινόμαστε καταναλωτές σε ένα και νεότερες ηλικίε. Επίσης αναπτύσσονται νέες καταναλωτικές συνήθειες όπως οι επιγραμμικές αγορές. Ε, ως εκ τούτου θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους κατανονισμούς και να ε, φροντίσουμε να ενημερώνονται οι καταναλωτές ακόμη και στα δημοτικά σχολεία τους ώστε η νέα γενιά να είναι ε, πιο υπεύθυνη ως προς καταναλωτικές τις συνήθειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει γενικότερη ενημέρωση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι θα αναβαθμιστεί η κατάστασή του, ε, διότι σε τι οφείλουν οδηγίε άμα δεν ξέρουμε πώ να τι χρησιμοποιήσουμε. Σα ευχαριστούμε, ο κύριο Χάρμπορ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής ε, και ως μέλος πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τον Κυριακό Τριανταφυλλίδη, διότι συνέχισε την καλή δουλειά που είχε κάνει η Εύα Πριτ Σβένσον. Είναι ατυχές ε, που μια τόσο φιλόδοξη και ευρύτατη έκθεση τελικά πρέπει να περιοριστεί ε, σε αυτήν την τόσο σύντομη συζήτηση, γιατί δεν προβλέπεται πλήρη συζήτηση για την έκθεση. Ε, παρόλα αυτά, Πιστεύω ότι απευθυνεί πραγματική έκκληση προ την Επίτροπο Ντάλ και θα ήθελα να σα καλωσορίσω εν παρόδο, ε, ούτως ώστε να είναι πιο φιλόδοξο σε σχέση με την πολιτική για την προστασία των καταναλωτών που τώρα εκπονεί. Ε, οι συντονιστέ των Επιτροπών ζήτησαν αυτή την έκθεση Ακριβώ για να τροφοδοτήσουμε αυτή τη διαδικασία, την εξέταση του ζητήματο. Όταν εξετάζει κανεί την έκθεση, εντοπεί ότι τώρα έχουμε μια ε, πολύ ρεαλιστική θέση. Έχουμε θέματα που αφορούν ε, τον κύριο Μπαρνιέ, τον κύριο κάνει την κυρία Ρέντινγκ ε, θέματα της ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δηλαδή, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόκληση στην οποία ε, καλείστε, Επίτροπε Ντάλη, να αντεπεξέλθετε και ευελπιστώ ότι θα προτείνετε μια ευρύτατη δέσμη μέτρων, ούτω ώστε να μα προσφέρει το πλαίσιο που χρειαζόμαστε για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για να προστατευθούν ικανοποιητικά, για να προχωρήσει στη συνέχεια με ουσιαστικό τρόπο η εσωτερική αγορά. Thank you, Mr. Harbour. Madame Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Εύα Μπριτ Σβένσον και τον συνάδελφο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη για την ε, δουλειά που έκαναν σχετικά με την εκπόνηση νέα στρατηγική ε, στον τομέα τη προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το τομέα να αποδώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ε, στι ανάγκε των καταναλωτών, κυρίω όταν μιλάμε για τι πιο ευάλωτε πληθυσμιακέ ομάδε μεσούσει τη σοβαρότατη χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει πολλά κράτη-μέλη. Πέρα από τι εκστρατείε ενημέρωση ελέγχου, δοκιμών των προϊόντων, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι όλε οι πληθυσμιακέ ομάδε, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκε, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, όλοι πρέπει να έχουν το επαρκές εισόδημα ώστε να έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά και υπηρεσίε, συγκεκριμένα ε, τρόφιμα αλλά και υπηρεσίε στον τομέα τομέα της υγείας, ε, της ενέργειας, ε, των ε, μεταφορών, της ευπρεπούς στέγης, ούτως ώστε να ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Ο Μπρικάδο, η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, όσον αφορά την ατζέντα και την προστασία των καταναλωτών. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα συνεκτικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκή προστασία των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παραπλανητική διαφήμιση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Ρουμανικές Εθνικές Αρχές για την Προστασία των Καταναλωτών ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα για να αλλάξουν την νομοθεσία στον τομέα αυτό τους ώστε να προστατεύσουν καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες στο χώρο της εκπαίδευσης και των ενημερωτικών εκστρατιών. Στη Ρουμανία για παράδειγμα υπάρχει ένας ετήσιος διαγωνισμός, εθνικός διαγωνισμός για την προστασία των καταναλωτών που διοργανώνεται από την Εθνική Αρχή και το Υπουργείο Παιδείας. Ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται τώρα στο ένατο έτος του και αφορά ανθρώπους και φοιτητές μεταξύ 6 και 18 και ο στόχος είναι εκπαιδευτικός. Ε, η έκθεση αυτή είναι αρκετά καλή, αλλά με εντυπωσιάζει πάντοτε το γεγονός πόσο αδιάφορο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναντι των ε, πολιτών, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Εμείς ε, λέμε ότι, λέμε ότι οι πολίτες ε, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας, αλλά στην πραγματικότητα ενισχύουμε τις δυνάμεις της αγοράς. Η προστασία των καταναλωτών είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχος αλλά πρόκειται για ευπαθείς ομάδες όπως τα παιδιά που χρήζουν προστασίας. Θα πρέπει να έχουμε μια πρόταση για απαγόρευση της διαφήμισης για τα παιδιά γιατί έχει δυσμενείς ε, επιπτώσεις ε, στα παιδιά. Οι διαφημίσεις αυτές αφορούν ήδη ένδυσης και παιχνίδια και δείχνουν πολύ γρήγορα, αποδεικνύουν κατά πόσο μια οικογένεια εύπορη ή όχι. Εμείς δεν θέλουμε ε, μια Ευρώπη των ε, αποκλεισμών ήδη στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό ε, θεωρώ ευκταίο να περάσουμε την εικόνα της κοινωνικής Ευρώπης. Ο τελευταίος ομιλητής θα μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασία των καταναλωτών που θα ψηφίσουμε αύριο λέει η κυρία Λεγκρίπ, βάζει κάποια ορόσημα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία θα θέλαμε να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προτείνει το, τη νέα ατζέντα για τους καταναλωτές αρχές του 2012. Ε, μεγαλύτερη ευθύνη των καταναλωτών, μεγαλύτερη ενημέρωση, να, να υπάρχουν ασφαλή προϊόντα για αυτούς θα πρέπει να εφαρμοστεί η, γρήγορα η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλοι να γνωρίζουν τι υποχρεώσει και τα δικαιώματά του. Αυτέ πρέπει να είναι οι προτεραιότητε για του εθνικού νομοθέτε και τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Αλλά και για τι επιχειρήσει, για τι επαγγελματικέ οργανώσει και τι οργανώσει των καταναλωτών. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε έναν βαθύ προβληματισμό για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των πληροφοριών, την πυκνότητα των πληροφοριών που χρειάζονται πραγματικά οι καταναλωτέ, τη χρήση που μπορούν να του κάνουν κατά τη διάρκεια τη αγορά του και το διοικητικό άχθο που η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών θα επισύρει για τις επιχειρήσεις. Επομένως, η βασική λέξη, λέξη κλειδί είναι ευθύνη των επιχειρήσεων, των ε, επιχειρηματιών, των παρόχων υπηρεσιών, αλλά και ευθύνη των καταναλωτών των ιδίων. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Επίτροπος Νταλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Σας ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ΙΜΚΟ και κυρίως τον εισηγητή, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, καθώς και την προηγούμενη εισηγήτρια, την κυρία Εύα Μπριτ Σβένσον, για την ε, έκθεση για μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασία των καταναλωτών. Καταλαβαίνω ότι η έκθεση είναι μια σειρά από συμβιβασμού και ίσω να μην αντιμετωπίζει, τουλάχιστον να μην αντιμετωπίζει πλήρω όλα τα θέματα που ορισμένοι από εσά θεωρείτε, ή ο καθένα από εσά θεωρείται πιο σημαντικά. Πάντω, το τελικό αποτέλεσμα τη ε, δουλειά σα είναι πολύ σημαντική συνεισφορά στη δουλειά και στο έργο τη Κομισιόν για την πολιτική ε, καταναλωτών. Έχει πολύ σημαντική σημαντικά στοιχεία για την πρόθεση των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Κυρίως, ε, καλωσορίζω πολύ την ε, σφαιρική προσέγγιση ε, που έχει αυτή η έκθεση για τους καταναλωτές. Μία επιτυχημένη πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο σε επίπεδο νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι πολυσχηδή. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση πολύ σωστά θέτει έμφαση στην ασφάλεια των καταναλωτών και για τα προϊόντα και για τα τρόφιμα. Τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ε, εξουσίας των καταναλωτών, της ε, παιδείας τους, των πληροφοριών που έχουν. Μιλάει ε, για την ανάγκη για μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την καινοτομία στο λιανεμπόριο και την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και με την παραπλανητική διαφήμιση. Μιλάει και για αυτά. Ε, μιλάει επίσης και για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών ε, και τις θέτει όλες αυτές ως προτεραιότητες. Μιλάει για την ανάγκη αποτελεσματικής ε, εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, τονίζει κάποια σημαντικά θέματα όπως βιώσιμη κατανάλωση, προστασία των επαθών καταναλωτών και πρόσβαση, προσπελασιμότητα. Αυτό το τρίγωνο επίσης δεν ξεχνάει και την ενέργεια, τα ψηφιακά και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επίσης υπήρχαν άλλες εκθέσεις. Ε, ε, επέρχεται μία έκθεση για τους ευάλωτους καταναλωτές και όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές οι εκθέσεις θα είναι πραγματική έμπνευση για την Κομισιόν, για τη μελλοντική πολιτική. Να σας πω ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ και εγώ θα παρουσιάσουμε την ατζέντα των καταναλωτών, θεματολόγια των καταναλωτών, το πρώτο εξάμεινο του επόμενου ε, έτους. Θα είναι μια πλήρης ε, ε, στρατηγική για τα επόμενα έτη. Μαζί με τα ορόσημα που θα τεθούν από το 2012 θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και θα βάλουμε του καταναλωτέ στο κέντρο τη εσωτερική αγορά. Αυτό το είπατε και εσεί, κ. Τραφιλίδη, στην έκθεσή σα. Η βασική αρχή θα είναι να δώσουμε δύναμη στου καταναλωτέ με την ευρία έννοια του όρου. Ε, ενίσχυση τη δύναμή του σημαίνει ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά οι καταναλωτέ στην αγορά και να τη χρησιμοποιήσουν προ όφελό του. Θα βάλουμε θέματα των καταναλωτών ε, στο χαρτοφυλάκιο τη κυρία Ρέντινγκ και φυσικά αυτά που είναι στο δικό μου, αλλά ε, μιλάμε και για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, ε, ψηφιακά θέματα, που είναι χαρτοφυλάκιο άλλων ε, επιτρόπων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Το θεματολόγιο των καταναλωτών θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις νέες προκλήσεις της πολιτικής αυτής θα πρέπει να έχουμε ε, πιο βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ ανάγκες ενός γυράσκοντος ε, πληθυσμού. Ε, τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, κοινωνική ένταξη, ευπαθείς καταναλωτές. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι συνάδουν αυτά που λέτε εσείς στην έκθεσή σας. Επίσης το θεματολόγιό μας θα έχει την φιλοδοξία να βασιστεί στην πρόοδο που έχει ήδη ε, σημειωθεί για την ε, υλοποίηση του ευρωπαϊκού ε, δικαστικού χώρου. Επομένως, οι δικαστές, τα νομικά επαγγέλματα θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη για να αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα. Η ατζέντα επίση θα βασιστεί σε εταιρικέ σχέσει, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουμε από κοινού του πόρου με βάση την αρχή doing more with less, κάνουμε περισσότερα με λιγότερα και αυτό σημαίνει εταιρικέ σχέσεις με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή και την ενημέρωση ε, με διαμέσους ε, της ε, οργανώσεις των καταναλωτών, με κέντρα ενημέρωση για τους καταναλωτές. Έχουμε ήδη συνεισφορέ από, από διάφορα δίκτυα συμβουλευτικά που λαμβάνουν υπόψη τα όσα λένε οι οργανώσεις καταναλωτών. Στις αρχές του 2012 θα οργανώσουμε και μια ακρόαση με τη, βοηθεία, τη επιτροπή της ΙΜΚΟ και συνεχίζουμε τις συζητήσεις για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Ως πρώτο βήμα ετοιμαζόμαστε ε, για μια ε, έκθεση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα θέματα των κατηνολωτών και τα οποία θέλουμε να τα εσωματώσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, από εσά. Την περασμένη εβδομάδα ε, υιοθετήσαμε ε, ένα πρόγραμμα ε, για τους καταναλωτές 2014-2020. Το συζητάμε τώρα στο... οι δημοσιονομικές αρχές. Έχουμε τέσσερις ε, τομείς δράσης. Καλύπτουμε όλα τα στοιχεία της πολιτικής καταναλωτών. Ε, με μεγάλη χαρά θέλω να σας πω ότι οι στόχοι αυτοί ε, συνάδουν με τις συστάσεις της εκθεσής σας. Η ασφάλεια των καταναλωτών, ε, προϊόντα, τρόφιμα και υπηρεσίες σωστές πληροφορίες και παιδεία, εκπαίδευση για τους καταναλωτές ώστε να καταλαβαίνουν ε, όλα αυτά τα πράγματα, ε, περισσότερα ένδικα μέσα στη διάθεση των καταναλωτών και τελευταίο εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τελευταίο αλλά σημαντικό. Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ε, ε, πολιτική κατανάλωση έχει ολοκληρωθεί. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι